Witam Państwa Συνεχίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με την επεξήγηση ψήφου. Γνωρίζω ότι το περιμένετε αυτό, περιμένετε αυτή τη στιγμή με ανυπομονησία. Εγώ αναλαμβάνω τώρα την Προεδρία και θέλω να ζητήσω από όσου παραμένουν στο ημικύκλιο, χωρίς όμως να σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τις επεξηγήσεις ψήφου, να αποχωρήσουν. Αν θέλετε να πάτε να φάτε στην καντίνα, στο εστιατόριο, πηγαίνετε ησύχω για να προχωρήσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Επεξηγήσεις ψήφου λοιπόν πρώτα απ' όλα για την έκθεση όσον αφορά την επισητιστική ασφάλεια. κυρία Μορβέ είναι η πρώτη.